μπορέσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες, οι αρχές, οι λιμένες να ε, προσαρμοστούν και κατόπιν να ξεκινήσει η εφαρμογή. Όταν ξεκινήσει η εφαρμογή, κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε Κάλλας, έχω ε, ένα συγκεκριμένο αίτημα. Ξεκινήσετε τώρα μια καμπάνια, μια εκστρατεία ενημέρωσης για τα δικαιώματα των επιβατών. Θα σας ζητήσω να να ξεκινήσετε σε 24 μήνες όταν τεθεί σε ισχύ ο κανονισμός για τα δικαιώματα των επιβατών ε, στη, στο θαλάσσιο τομέα να ξεκινήσετε μια εξίσου ωραία ε, καμπάνια και για τον τομέα αυτό. Το αξίζει νομίζω αυτό ο Ευρωπαίος πολίτης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ολοκληρώνεται η συζήτηση. Η ψηφοφορία θα λάβει χώρα αύριο στις 12. Now we pass, we move. Και τώρα Πάμε. Στη σύσταση για δεύτερη ανάγνωση του κειμένου της κυρίας Γένσεν εφή συστήματα μεταφορών στον τομέα των οδικών μεταφορών και διεπαφή με άλλους τρόπους ε, μεταφορών. Θα δώσω το λόγο στην Αν Γένσεν που είναι η συγγήτρια για τέσσερα λεπτά έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όσον αφορά τα ευφυή e e συστήματα μεταφορών, ε, για τι πράγμα μιλάμε. Πρόκειται για όλα τα συστήματα πληροφοριών, πληροφορικής που μπορούν να διευκολύνουν τις μεταφορές, να γίνουν πιο αποτελεσματικά και να σέβονται το περιβάλλον τα μεταφορικά μέσα. Το GPS που χρησιμοποιούμε παραδείγματο χάρη ε, μπορεί να βοηθά και στην καταβολή ε, των ε, διοδίων, αλλά υπάρχουν και άλλα συστήματα τα οποία προετοιμάζονται, διάφορα συστήματα τα οποία θα μας επιτρέπουν να έχουμε καλύτερες πληροφορίες όσον αφορά το χρόνο που χρειάζεται αυτοκίνητα να διανύσουν μια απόσταση, αν υπάρχουν ουρές, αν έχουν συμβεί ατυχήματα, έχουν αυτόματο σύστημα που θα μπορεί να καλεί το κέντρο όταν συμβαίνει ένα ατύχημα για να φτάνει και πιο γρήγορα η βοήθεια. Με αυτή την έκθεση από την αρχή είχα διάφορες απογοητεύσεις. Διερωτήθηκα καταρχήν τι είναι αυτό το FES μεταφορικό σύστημα, διότι καλύπτει ένα ευρύ φάσμα και ήθελα να δω και ποιες δυνατότητες υπάρχουν όσον αφορά τα συστήματα και απογοητεύτηκα όσο μελετούσα το θέμα και λυπήθηκα διότι δεν είχαμε ήδη αυτά τα συστήματα. Όταν είναι κανείς ε, σε ένα μποτιλιάρισμα δεν μπορεί και χάνει το αεροπλάνο του ε, είναι πρόβλημα αυτό και τα πράγματα θα κυλούσαν πολύ πιο ομαλά αν υπήρχαν και άλλες πληροφορίες. Γιατί δεν έχουμε μέχρι τώρα αυτά τα συστήματα. Οι εμπειρογνώμονες Ευρωπαϊκής Επιτροπής μας είπαν ότι έλειπαν προδιαγραφές και πρότυπα που θα επέτρεπαν την προώθηση της χρήσης αυτών των εφιών συστημάτων, την παραγωγή τους και να είναι πιο εύκολο να εφαρμόζονται σε όλες τις χώρες. Να πηγαίνει ένα φορτηγό από τον Κέντρο στο Παλέρμο χωρίς να υπάρχει πρόβλημα, να μπορεί να επικοινωνεί με όλα τα συστήματα που υπάρχουν. Χωρίς η διαδρομή να εμποδίζεται από έλλειψη δελειτουργικότητας. Θα πρέπει να καθοριστούν προδιαγραφές σε τέσσερις τομείς και θα πρέπει να προβλέψουμε και έξι σχέδια δράσης, έξι άξονες δράσης. Θα πρέπει να δίδονται πληροφορίες όσον αφορά την ασφάλεια, να δίδονται πληροφορίες όσον αφορά την οδική ασφάλεια εν γέννη, να εξασφαλίζεται η εφαρμογή του e-call και κάτι πάρα πολύ σημαντικό, να μπορούν οι οδηγοί να έχουν τις πληροφορίες όσον αφορά τα σημεία στάθμευσης που είναι ασφαλή και να μπορούν εκ των προτέρων να κρατούν κάποια θέση και να είναι λιγότερο αγχωμένοι όταν οδηγούν τα φορτηγά και χρειάζονται ανάπαυση. Ε, η δουλειά που κάναμε είναι αυτή. Λοιπόν, αντιμετωπίσαμε την πρακτική εφαρμογή των συστημάτων αυτών και είχαμε συμφωνήσει στο Κοινοβούλιο ότι θα πρέπει να καθορίσουμε τους τομείς εκείνους που χρειάζονται ειδικέ κοινέ προδιαγραφές. Το Συμβούλιο όμως τελικά δεν προσήγγισε τις προτάσεις μας, κυρίως όσον αφορά την πρακτική εφαρμογή όλων αυτών των μέτρων. Και προβλέψαμε δύο φάσεις. Πρώτα απ' όλα να καθοριστούν προδιαγραφές και δεύτερον θα πρέπει να εξεταστεί το πώς θα εφαρμοστούν αυτές. Θα ήθελα να πω ότι υπήρξε καλή συνεργασία θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Τικάου, τον κύριο Κόκ και την κυρία Πόλς, όλος ιδιαίτερος. Ε, νομίζω ότι η συνεργασία μας ήταν πολύ στενή και θα ήθελα να ευχαριστήσω και ιδιαίτερα τη Σουηδική Προεδρία που κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες ούτως ώστε η πρόταση αυτή του Κοινοβουλίου να μπορεί να περάσει το τελικό κείμενο του Συμβουλίου. Και μετά ένα μεγάλο ευχαριστώ επίσης την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματικά βοήθησε να γεννηθεί αυτό το κείμενο και συνέβαλε ε, στο να καταλήξουμε σε αυτή την κοινή συμφωνία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Γένσεν. Και τώρα το λόγο τον δίνουμε στον Επίτροπο, τον κύριο Σιμ Κάλλας. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρόεδρε Αξιότιμη Κυρίε και κύριοι βουλευτέ, θέλω να ευχαριστώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα την κυρία Γένσεν, την εισηγήτρια για τα εφή συστήματα μεταφορών, αλλά και όλου του για το εξαίρετο έργο του και την συνεχή του στράτευση στην στήριξη των προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για τη διαδικασία αυτή που οδηγεί στην οδηγία. Η δεύτερη ανάγνωση λοιπόν η φινομοθετική πρόταση επί του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με φέρει ενωπιόν σα για να επιβεβαιώσω για άλλη μια φορά με απερίφραστου κατά των όρου την τεράστια πολιτική τη σημασία και κάθε είδου ε, συνθήκε μεταφορών εφιών, ηλεκτρονικών ε, σύστημα παρακολούθησης ή πληρωμής διοδίων διευκολύνουν τον επιβάτη, μειώνουν το χρόνο της ε, μεταφοράς και να ισχύουν την ασφάλεια. Έχει προσπαθήσει η Επιτροπή διαρκώς να προαγάγει τις ε, μεθόδους ή τις λύσεις που προσφέρει η νέα τεχνολογία. Στις οδικές μεταφορές όμως πρόοδος ήταν πολύ βραδύτερη από ό,τι σε άλλους, τρόπους μεταφορών και πολλές φορές μάλιστα κατακαιρματισμένη συμφωνίες, τυποποίηση που προσπαθήσαμε να αναπτύξουμε δεν προσέφεραν επαρκή πρόοδο ως προς την ανάπτυξη και χρήση τέτοιου είδους συστημάτων. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβάλλει ένα πρόγραμμα δράσεως και πρόταση για οδηγία πλαίσιο ως προς την ανάπτυξη εφιών συστημάτων μεταφορών στις οδικές μεταφορών, μεταφορές και, τις, ε, και τη διεπαφή με άλλες μορφές μεταφορών, με τύπους μεταφορών. έτσι και με τις διαπραγματεύσεις που έγινε με το Συμβούλιο βλέπουμε μια πρόταση αρκετά ισορροπημένη και βλέπουμε ότι λαμβάνονται υπόψη οι τα ιδιαίτερα σημεία που επιθυμούσε η Επιτροπή να προχωρήσουν. Ευχαριστώ ιδιαίτερα την κυρία Γέννης. Είμαι πολύ ικανοποιημένο από τις, προσπα... από τις προτάσεις που υιοθέτησε στις 22 Ιουνίου η Επιτροπή των Μεταφορών και προσβλέπω στην έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της οδηγίας ε, αυτή στην αυριανή σα συνεδρίαση προχωρούμε ταχύτατα μόλις εγκριθεί η οδηγία στην εφαρμογή της, στην συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς του δυτικού και δημοσίου τομέα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αντιπρόεδρε. Το λόγο έχει ο συνάδελφος Δίτερ Κοχ για 1,5 λεπτό. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η οδηγία για την εισαγωγή και χρήση ευφυών συστημάτων στις οδικές μεταφορές και ιδιαίτερα των σημείων συνάντησης με τους άλλους τύπους των μεταφορών έχει τεράστια σημασία. Θα ήθελα να μιλήσω δηλαδή για την εκκίνηση μιας νέας εποχής στις οδικές μεταφορές. Έχουμε να κάνουμε με ένα πρόγραμμα δράσης μας που έχει υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το οποίο εξασφαλίζει την εισαγωγή νέων ε, υποδομών, νέων τεχνολογιών για τα οχήματα και τα οδικά μας συστήματα. Δεν είναι σαφές όμως πότε θα καταστεί υποχρεωτική η εισαγωγή αυτών των νέων ευφυών συστημάτων. Θα ήθελα να υπάρχει κάποια συγκεκριμένη προθεσμία. Δεύτερον, οι μεταφορές θα είναι πιο καθαρές, πιο αποτελεσματικές, πιο ασφαλείς. Και η διαλειτουργικότητα αλλά και η διασύνδεση των διαφόρων μέσων μεταφοράς θα πρέπει να εξασφαλιστούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Ήψιστο ε, ποσοστό επίσης ε, ποιότητας, υποδομών και υπηρεσίας τόσο για τον ιδιώτη όσο και για την επιχείρηση πρέπει να επιδιώξουμε όλοι. Η έκθεση λοιπόν πιστεύω συμβάλλει σημαντικά στην πρόοδο και το μέλλον των οδικών μεταφορών και την εξυπηρέτηση των στόχων του 2020. Με τα νέα αλλά και τα εφιστάμενα συστήματα το Κοινοβούλιο πιστεύω καταβάλει ιδιαίτερες προσπάθειες για να συμβάλλει προς το στόχο αυτό. Το ΕΛΚ ιδιαίτερος δίνει έμφαση στην έννοια του e-call και των άλλων ηλεκτρονικών συστημάτων ενημέρωσης αλλά και κράτησης έτσι ώστε να έχουμε την ευρύτερη δυνατή κάλυψη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση το ταχύτερο δυνατό. Ευχαριστώ κύριε Κόχ. Το λόγο τώρα έχει η κυρία Σίλβια Ντριάννα Τικάου. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, η υιοθέτηση μιας οδηγίας πλαισίου για την εφαρμογή των ευφυών συστημάτων ε, μεταφορών αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό βήμα μπρο για να εξασφαλίσουμε αύξηση της ασφάλειας στις μεταφορές. Θέλω να ευχαριστήσω την ομάδα των εισηγητών διότι διεύρυνε το πεδίο εφαρμογή τη οδηγία ε, από τις οδικέ μεταφορές περιλαμβάνοντας και τις επαφές με άλλα μέσα μεταφορών. Τα, τα ευφύ αυτά συστήματα θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τέτοιο τρόπο ώστε ε, και οι οδικέ μεταφορέ και οι διαπαφέ του, και συμπεριλαμβανομένων των οδικών μεταφορών να καλύπτονται αφορώντα ταυτόχρονα και άλλα μέσα μεταφορών. Το Κοινοβούλιο από την πρώτη ανάγνωση είχε ζητήσει ένα ελάχιστο επίπεδο για τι εφαρμογέ των, των συστημάτων μεταφορών και αυστηρέ ε, προδιαγραφέ για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η οδηγία περιλαμβάνει τέσσερι βασικού ε, κλάδους προτεραιότητες στους οποίους πρέπει να θεσπίσει κοινού κανόνες και ελάχιστες προδιαγραφές η Επιτροπή. Η Επιτροπή ανέλαβε τη δέσμευση να εγκρίνει εντάχει τους, ε, τις ειδικές προδιαγραφές μέσα σε ένα χρονοδιάγραμμα που θα ολοκληρωθεί το 2014 επιτρέποντας τη χρονιά εκείνη να μπουν στην Ευρώπη σε λειτουργία τα συστήματα αυτά. Και Επίσης, το 2013 θα πρέπει να υπάρχει online ενημέρωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τις ε, ε, για την κυκλοφορία καθώς και το 2012 γενικές πληροφορίες πληροφοριών σε δωρεά, με δωρεάν παροχή για τις οδικές μεταφορές. Επίσης, το 2012 δεσμεύτηκε να υπάρχει ένα σύστημα διαλειτουργικότητας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και την ίδια χρονιά και το 2013 η εισαγωγή ενός συστήματος πληροφόρησης που θα επιτά ε, εξασφαλίζονται θέσεις, θέσεις για τα φωτιγά. Οι διατάξεις αυτές πρέπει να ενημερωθούν με τις νέες διατάξεις της ε, Λισαβόνας στην επιτροπολογία και την χορήγηση ε, πράξεων στην Επιτροπή. Πιστεύω ότι ο τρόπος αυτός θα βελτιώσει τις μεταφορές και ότι τα κράτη-μέλη και η Επιτροπή θα παράσχουν τα επαρκή κονδύλια για τη λειτουργία του συστήματος. Ευχαριστούμε κύριε Τικάου. Η κυρία Μέσνερ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κόχ ο κύριος Κόχ έχει δίκαιο. Πρόκειται για την εκκίνηση μιας νέας εποχής οδικές μεταφορές. Αυτό μας προσφέρουν οι συστήματα. Έχω δει πρόσφατα να συνομιλούν μεταξύ τους φορτηγά. Απίστευτο, αλλά αληθινό. Αυτά μας φέρνει τεχνολογία και το μέλλον. Μπορεί ένα φορτηγό να αναγνωρίσει χάρη σε ένα μηχάνημα, ένα άλλο, είναι ενημερώσει αν υπάρχει μπροστά εμπόδιο, αν υπάρχει πεζό στο δρόμο, να βοηθήσει έτσι ώστε εγκαίρως να φρενάρει ο οδηγός και να αποφευχθεί το ατύχημα. Η κυρία Γένσεν λοιπόν έχει καταβάλει ιδιαίτερη προσπάθεια να καταγράψει με ευρύτερη, ευρύτερη επισκόπηση όλες τις δυνατότητες που προσφέρει σήμερα η τεχνολογία αλλά και που θα έχουμε και στο μέλλον για να βελτιώσουμε την ασφάλεια των οδικών μας μεταφορών, για να έχουμε πιο ασφαλείς δρόμους και καλύτερες μεταφορές. Εγώ στη Γερμανία όπου μένω κοντά στο Ανόβερο έχουμε μπορέσει να χρησιμοποιήσουμε τεχνολογία αυτή για να παρακολουθήσουμε την βέλτιστη, για να εξασφαλίσουμε τη βέλτιστη ταχύτητα των οχημάτων, δηλαδή το, με τι ταχύτητα πρέπει να τρέχουν τα αυτοκίνητα έτσι ώστε να έχουμε και καλύτερη ροή κυκλοφορία, αλλά και λιγότερη μόλυνση. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μπρέπολ, έχει το λόγο για ένα λεπτό. Και μισό. Ε, ναι, λέει κυρία Μπρέπολς, ανάμιση λεπτό. Ευχαριστώ Προέδρε. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής διότι επιτέλους έχουμε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για τα ευφυή e συστήματα μεταφορών, όπως είπαν ήδη οι συνάδελφοι, ήταν δύσκολα τα πράγματα, δύσκολο να πετύχουμε το αποτέλεσμα. Χάρη όμως στην αφοσίωση και στις άοκνες προσπάθειες της συναδέλφου μας της κυρίας Γένσεν, μετά από μακρές δυσκολότατες διαπραγματεύσεις μπορούμε επιτέλους να καταλήξουμε αυτά τα αποτελέσματα. Μεγάλο ευχαριστώ κυρία Γένσεν. Βλέποντας τα προβλήματα της ρήπανση, τα προβλήματα της κυκλοφοριακής συμφόρηση δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε την σημασία της πρωτοβουλίας. Είναι σημαντικό να βρούμε καινοτόμε λύσεις. Και η ευρωπαϊκή προσέγγιση είναι ιδιαίτερα σημαντική, διότι οι δυνατότητες των εφιών συστημάτων δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν παρά μόνο να εισαχθούν ε, ομοιόμορφα τα μέτρα. Δεν μπορούμε να τα εφαρμόσουμε κατακαιρματισμένα. Χρειάζεται συντονισμένη ανάπτυξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτή είναι μια πρώτη φάση πολύ σημαντική όμως. Θα πρέπει όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη τα επόμενα χρόνια να παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς την εφαρμογή των τραφόρων δράσεων που έχουν προτεραιότητα. Ήδη έχουμε μείνει πίσω κατά ένα εξάμεινο συγκρίση με το χρονοδιάγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λόγω των συζητήσεων όσον αφορά την εφαρμογή αυτών των ανατεθ... ανατεθεμένων πράξεων, εκχωρουμένων πράξεων θα πρέπει να φροντίσουμε οι προβλεπόμενες υπηρεσίες να είναι αρκετά εύχριστες για τους διάφορους χρήστες και χαιρόμαστε διότι προβλέπονται κάποιες διατάξεις για τους χρήστες που είναι ευάλωτοι. Νομίζω ότι θα πρέπει να προσέξουμε όλος ιδιαίτερως αυτή την κατάσταση διότι θέλουμε να πετύχουμε ε, υπηρεσίες ποιότητας για όλους. Ευχαριστώ. Η κυρία Άννα Ρόσμπαχ έχει το λόγο για μισή λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στο παρμπρί αυτοκινήτου μου υπάρχει μια συσκευή που επιτρέπει να καταγράφεται η διέλευσή μου από τα διόδια. Και θα ήθελα να μπορεί να λειτουργεί το ίδιο σύστημα και σε γειτονική χώρα. Θα ήταν πάρα πολύ ευχάριστο αυτό, διότι έτσι θα μπορούσα εύκολα να ταξιδεύω σε όλη την Ευρώπη. Και εκεί θέλει να καταλήξουμε κυρία Γένσεν υπέρ όλων εκείνων που ταξιδεύουν πολύ στους ευρωπαϊκούς αυτοκινητόδρομους. Ευχαριστώ, Αν, για την δουλειά που έκανες στα πλαίσια της προσπάθειας που καταβάλλεται σε αυτή την οδηγία. Αυτή η οδηγία περιέχει διάφορα συγκεκριμένα στοιχεία τεχνικής φύσεως και δεν μπορώ παρά να ενθαρρύνω την κίνηση αυτή, την προσέγγιση αυτή για την κατάρτιση προδιαγραφών και την υλοποίηση της νομοθεσίας είναι ένα θέμα που συζητήθηκε, οδήγησε διάφορες προτάσεις ε, προτάσεις που είναι πολύ σημαντικές για τους οδηγούς των φορτηγών. Χωρίς αυτούς θα αμφισβητεί το ίδιο ύπαρξη Ευρωπαϊκής Ενώσεως χωρίς τους οδηγούς των φορτηγών. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις καλές προθέσεις που είναι στη βάση των προτάσεων αυτών. Ε, το Συμβούλιο δεν συμφωνεί απόλυτα με τη δική μας προσέγγιση, αλλά θα πρέπει να προχωρήσουμε βήμα-βήμα και θα πρέπει επίσης να επιδείξουμε πολιτική βούληση και για άλλες μεταφορικές μεθόδους όπως και τους σιδεδρόμους. Η κυρία, ευχαριστώ κύριε Ρόσμπαχ, για 1,5 λεπτό έχει το λόγο ο κύριος Κουμουτσάκος. Γιώργος. Κύριος Γιώργος Κουμουτσάκος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η εξάπλωση των ευφυών συστημάτων μεταφορών στις οδικές μεταφορές αλλά και στη λειτουργική του σχέση με τους άλλους τρόπους μεταφοράς είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα. είναι μια πραγματική πρόκληση για την ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών και ορθώ προηγούμενοι συνάδελφοι μίλησαν για μια νέα εποχή στι μεταφορέ. η ευρύτατη δυνατή εφαρμογή των ευφυών συστημάτων μεταφορών θα συμβάλλει πρώτον σε πιο αποτελεσματικέ πιο σταθερέ και πιο ασφαλεί μεταφορέ και δεύτερον στην επίτευξη του στόχου για καθαρότερε και φιλικότερε στο περιβάλλον μεταφορέ πιστεύω λοιπόν κύριε πρόεδρε ότι η έγκριση της οδηγίας πλαίσιο για τα ευφυή e e συστήματα μεταφορών θα είναι μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για όλους τους ευρωπαίους πολίτες και αυτό γιατί έως τώρα η εθελοντική προσέγγιση δεν λειτουργήσε καθόλου ικανοποιητικά. χρειαζόμαστε και όλοι συμφωνούμε σε αυτό ένα ελάχιστο επίπεδο τυποποίησης εάν θέλουμε να δούμε σε σύντομο χρονικό διάστημα τη χρησιμοποίηση αυτών των συστημάτων στα ταξίδια και τις μετακινήσεις μας και όπως η εισηγήτριά μα, η κυρία Γένσεν την οποία συγχαίρω πιστεύω ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε και να εγκρίνουμε αύριο προκειμένου ε, να επιβεβαιώσουμε άλλωστε ότι προηγήθηκε μια μακρά σκληρή διαπραγμάτευση που κράτησε μάλιστα έω πριν ε, λίγο καιρό και πρέπει τώρα να προχωρήσουμε. το τελευταίο που θα χρειαζόμασταν θα ήταν μια νέα αλλά αχρίαστη καθυστέρηση τη όλη διαδικασία και πάλι συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. ευχαριστώ πολύ κύριε πρόεδρε. Ευχαριστώ συνάδελφε. Το λόγο έχει η κυρία Γιάλα Σέντερ. 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και εγώ να συγχαρώ την κυρία Γένσεν γιατί πραγματικά πάλεψε για την πρόθεση αυτών των ευφυών συστημάτων μεταφορών στις οδικές μεταφορές για να πετύχει και εναρμόνιση και ε, συμβατότητα κυρίως. Αυτές τις ημέρες διάβασα πώς η SNCB στις Βρυξέλλες ε, κατόρθωσε να παράσχει στους οδηγούς ε, online ενημέρωση για την κυκλοφορία για να μπορέσουν να ε, τους επιτρέψει επαρκή χρόνο για την διαλειτουργικότητα κάτι που θα είναι μια βασική διάσταση των υπηρεσιών του μέλλοντος τόσο ώστε να μπορέσουν οι υπηρεσίες αυτές να προχωρήσουν με θεματικό τρόπο σε όλη την Ευρώπη. Αυτό απαιτεί όχι μόνο διάλογο αλλά και διασυνοριακό διάλογο στις οδικές μεταφορές που είναι μια βασική διάσταση της, της οδικής ασφάλειας. Ιδίως διότι θα είναι αναγκαίο να επεκταθεί το e-call σε όλη την Ευρώπη ε, ούτω ώστε να καλύψει όχι μόνο τις ευρωπαϊκές υποδομές αλλά και παραπέρα ιδίω για τα ε, οχήματα αγροτικής χρήσης σε περιοχές όπως την δική μου πολύ συχνά υπάρχουν ατυχήματα και ε, ο οδηγός ε, ε, πεθαίνει διότι δεν μπόρεσε να φτάσει έγκαιρα ή να φτάσουν έγκαιρα οι πρώτες βοήθειες. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι πολύ χρήσιμο να έχουμε τις ζώνες ασφαλούς στάθμευσης των μεγάλων οχημάτων που θα έπρεπε να επεκταθούν στο μέλλον όλο ένα και περισσότερο στην Ευρώπη και το μόνο που θα έλεγα είναι να μπορέσει το Γαλιλαίο να γίνει πλατφόρμα για τέτοιες υπηρεσίες. Αυτό θα ήταν πραγματικά το ιδεώδες. Ελπίζω ότι θα το πετύχουν αυτό ο κύριος Κάλλας και ο κύριος Σταγιάννη, ούτως ώστε το σύστημα των ευφυών συστημάτων μεταφορών να είναι το σύστημα του μέλλοντος. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Ο κύριος Ρώση έχει το λόγο για ένα λεπτό. Αξιότιμοι συνάδελφοι, πρόεδρε, καλύτερη διαχείριση τη μεταφορά εμπορευμάτων και μεγαλύτερη ασφάλεια οδική είναι δύο σημαντικέ πτυχέ στα πλαίσια τη δημιουργία ενό συστήματο ε, φιών μεταφορών. Στόχο να δημιουργήσουμε ένα συντονισμένο και ολοκληρωμένο σύστημα που θα εγγυάται μια συνέχεια των υπαρχή υπηρεσιών, διαχείριση τη κυκλοφορία, τη μεταφορά των εμπορευμάτων στου μακρύ αυτοκινητόδρομου ε, θα πρέπει θα έχει και συνέπειε οικονομικέ. Ε, κοστίζουν τα σημεία διαπαφή όσον αφορά κυκλοφορία και θα μπορούσε να επιληθεί το πρόβλημα μέσω τυποποίηση των διαφόρων συστημάτων και να έχουμε ολοκληρωμένο σύστημα πληροφορική. Αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα, συνέχεια, διαλειτουργικότητα είναι οι βασικέ επί των οποίων θα πρέπει ε, να εδραιωθούν οι προσπάθειε μα. Χρειάζεται σωστή αξιολόγηση των χαρακτηριστικών των περιφερειακών και των συνθήκων τη κυκλοφορία, των διαφόρων σημείων διαπαφή μεταξύ των διαφόρων μεθόδων μεταφορών μέσω μια εφαρμογή πραγματικά ε, αποτελεσματικού συστήματο. Χρειάζεται μια σειρά αξιολογήσεων του πώ αντιδρά σε στιγμέ κρίσιμες το σύστημα θα έπρεπε η Επιτροπή που δημιουργεί η οδηγία να μπορεί να συνομιλεί με την τοπική αυτοδιοίκηση για να μετρηθεί το σύστημα, ώστε να υπάρχει ταχεία και αποδοτική ανταπόκριση αν υπάρχουν διάφορα προβλήματα που συνδέονται συνδέονται με Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Ρώση. Και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Κώσα για 1,5 λεπτό. Η κυρία Κώσα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κώσα μάλλον. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να καλωσορίσω την παρέμβαση αυτή για τα μέτρα αυτά για τα εφή συστήματα μεταφορών γιατί υποστηρίζουν, ε, βοηθούν τον κόσμο ε, να ζήσει πιο εύκολα, θα ήθελα να υπογραμμίσω κάποια πράγματα. Πρώτα απ' όλα, είδαμε και στα δικαιώματα των επιβατών ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν αφοσιωθεί, σε, έχουν επιδοθεί σε μια προσπάθεια για να υποστηρίξουν τα άτομα με αναπηρία. Αλλά στο σύστημα αυτό επίσης θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στα άτομα με αναπηρίες και όταν τα συστήματα θα εισαχθούν και θα αναπτυχθούν, αυτή η πτυχή θα πρέπει συνεχώς να λαμβάνεται υπόψη και να εστιαζόμαστε επ' αυτών. Όσον αφορά την επικοινωνία και την ανταλλαγή πληροφοριών, εκεί θα πρέπει να έρθουν τα εμπόδια, θα πρέπει να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που έχουν αναπηρίες. Ε, ξέρουμε ότι λείπουν και κάποιες αξιολογήσεις αντικτύπου. Δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το κόστος εισαγωγής αυτού του συστήματος. Θα ήθελα να ζητήσω λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερους πόρους για αυτό το σκοπό, ώστε να γνωρίζουμε κατά πόσο στις χώρες Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης ε, μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό το κόστος και να καλυφθεί. Τώρα περνάμε στη δικασία Catch the Eye. Δίνω το λόγο στον κύριο Μαρινέσκου. Ε, ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η δημιουργία ενός ενιαίου πλαισίου χρήσης, συντονισμένης χρήσης των ευφυών συστημάτων μεταφορών αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την, τον εξυγχρονισμό των μεταφορών και υποχρεώνει το κράτη-μέλη να εξασφαλίσουν την υλοποίηση και εφαρμογή των συστημάτων αυτών με ε, διαλειτουργικό τρόπο. Ως εισηγητής για τους ευρωπαϊκούς διαδρόμους εμπορικών μεταφορών πιστεύω ότι τα, τα αυτά συστήματα είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για τη διαχείριση ιδίω των μεταφορών και γι' αυτό χρειάζεται να υπάρξει αμοιβαία αναγνώριση της έγκρισης τύπου και των προδιαγραφών σε εθνικό επίπεδο για όλους τους εξοπλισμούς και τα προγράμματα και σεβασμός των προγραμμάτων ανάπτυξης των, συστημάτων ε, ETMES, ούτως ώστε να προσαρμοστούν στις απαιτήσει των νέων συστημάτων. Ήδη το ότι έχουμε προχωρήσει είναι θετικό και πρέπει να αποφύγουμε να υπάρχουν ε, διακοπές γεωγραφικού χαρακτήρα. Ο κύριος Κέλλη έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι θα ήταν ανόητο να αντιταχθεί κανείς σε ευφυείς προτάσεις. Και σίγουρα τα ευφυείς συστήματα μεταφορών δεν μπορούν να βρουν αντίπαλο, θα πρέπει να είναι πρόσδεκτα. Ε, συγχαίρω την κυρία Γέντσεν και τον κύριο Κάλλας που υπογραμμίζουν τα θετικά στοιχεία. Θέλουμε οι μεταφορές να είναι φιλικές προς το περιβάλλον, να θέλουμε να αυξηθεί η οδική ασφάλεια. Θέλουμε να υπάρχει σωστή ε, στάθμευση, να μπορούμε να έχουμε και ενημέρωση όσον αφορά τι καιρικέ συνθήκε κλπ. Είναι πολύ σημαντικό. Όσον αφορά την οδική ασφάλεια, θα ήθελα να τονιστεί το ότι οι... τι συνέπειε έχουν οι αργοί οδηγοί, αυτοί που οδηγούν αργά στα ατυχήματα. Όλοι τονίζουν την ταχύτητα και αυτή συμβάλλει στα ατυχήματα πολύ. Ε, θα ήθελα να, πω στην ευφυή κυρία Γένσεν ότι την ευχαριστώ πολύ που βοηθά η χρήση των δρόμων να γίνει αποφελής ε, για όλους τους χρήστες, είτε είναι ανόητοι, είτε είναι έξυπνοι, είτε είναι ευφύης. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κάντζα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πιστεύω ότι είναι πολύ χρήσιμο ο ορισμό αυτών των προδιαγραφών για την ανάπτυξη συντονισμένη των συστημάτων και των διαφόρων εφαρμογών ITS στα δίκτυα των μεταφορών και στι αερομεταφορέ. Θα ήθελα να υπογραμμίσω όμω δύο πράγματα όσον αφορά την ασφάλεια. Το πρώτο είναι θα πρέπει να επιμείνουμε πολύ επί των ασφαλών χώρων σταθμέσεω για τα φορτηγά. Και δεύτερον, για τι οδικέ μεταφορέ. Και όταν μιλάμε για ασφάλεια και οι οδηγοί στου οδηγού φτάνουν πάρα πολλέ πληροφορίε που όλο και αυξάνονται και κατακλείζονται, θα πρέπει να προσέχουμε διότι θα πρέπει να κάνει τα πάντα εκτός από τον οδηγεί οδηγός. Ε, σήμερα αυτό είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό και αυτή η πτυχή είναι κάτι που θέλω να θέσω προς την κυρία Γένσεν διότι ε, νομίζω ότι από τη μια πλευρά Υπάρχει αυτή η βούληση. Από την άλλη όμως θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί να φροντίσουμε ούτω ώστε να σκέφτεται ο οδηγό ότι και να έχει και το νου του και στην οδήγηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δίνω το λόγο στον κύριο Όμπερμαϊερ. Πρόεδρε, Η ασφάλεια οδικέ οδικές μεταφορές είναι εκ των χρόνων κανεφόρο για μια ε, για ποιοτικές μεταφορές και θα ήθελα ιδιαίτερος να υπογραμμίσω ε, ε, την ανάγκη να μην κυκλοφορούν στους ευρωπαϊκούς δρόμους τα τεράστια, πολύ μεγάλα φορτηγά τα οποία κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή. Γιατί σε περίπτωση ατυχήματος έχουν τεράστιες ε, συνέπειες για, την, ε, για ολόκληρο το περιβάλλον, ιδιαίτερα όπως είδαμε στην περίπτωση του ατυχήματος του Μπρούνερ. Και επίσης θα πρέπει να μεριμνήσουμε για τις συνθήκες, για, τον εξοπλισμό ασφάλειας θα μπορούσε να εισαχθεί και στα αγωνιστικά αυτοκίνητα, ο οποίο δεν κοστίζει παραπάνω από 50 100 ευρώ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Ροντζούλη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι Ευρωπαίοι πολίτε ετοιμάζονται αυτή τη στιγμή να φύγουν για τι ε, καλοκαιρινές διακοπέ. Δυστυχώ, όπως κάθε χρόνο, θα πρέπει να αντιμετωπίσουν ακυρώσει πτήσεων, ε, κυκλοφοριακή συμφόρηση, Κατάστασει που είναι ε, ακραίες αλλά τις οποίες έχουμε πλέον ε, συνηθίσει. Την περασμένη εβδομάδα υπήρξε δέσμευση της Επιτροπής να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Η κίνηση μιας καμπάνιας ενημέρωση για τα δικαιώματα των επιβατών αποτελεί ένα χρήσιμο αλλά όχι επαρκές μέσο για να αποφύγουμε τέτοια προβλήματα. Πολύ συχνά τα δικαιώματα των ταξιδιωτών παρα, παραγνωρίζονται και για να πάρουν αποζημίωση μπορεί να χρειαστεί να περιμένουν μήνες και χρόνια. Η ενημέρωση, η γνωστοποίηση των δικαιωμάτων κάποιου είναι σημαντικό. Αλλά πολύ σημαντικότερο είναι η υλοποίηση στην Ευρώπη, σε ολόκληρη Ευρώπη, συγκεκριμένων μέτρων για ε, γεγονότα που συνήθως είναι γνωστά και μπορούν να αποφευκούν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ροντσούλη. Κύριος Κάλλας έχει το λόγο τώρα, ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κυρίε και κύριοι βουλευτές, θα ήθελα για άλλη μια φορά να ευχαριστώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την κυρία Γιάννησαν ιδιαίτερω για την πολύ καλή δουλειά στην νομοθετική διαδικασία που οδηγεί στην έγκριση ενό συστήματο εφιών οδικών μεταφορών. Με δημονία περιμένω και την πολύ σημαντική δουλειά που έχουμε μας περιμένει στην εφαρμογή της οδηγίας αυτής. Είμαστε βεβαίως ε, έτοιμοι να αξιοποιήσουμε τις εξουσίες που έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσα στα στην επόμενη επταετία για την εφαρμογή των συγκεκριμένων ε, διατάξεων εφαρμογής σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Η κυρία Αν Γένσεν έχει τώρα το λόγο, η σύντρια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τις παρατηρήσεις τους. Πιστεύω ότι η συζήτηση αποδεικνύει ότι υπάρχει ευρεία συνένεση και αποδοχή, αλλά και πολλές προσδοκίες με το σχέδιο αυτό. Θέλω να ευχαριστήσω ιδίως τον κύριο Επίτροπο για την υπόσχεση που έδωσε να ε, αγωνιστεί για να υπάρξουν συγκεκριμένα αποτελέσματα και τη δέσμευσή του να αναλάβει ευθύνε για την συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Η Επιτροπή δεσμεύθηκε επιπλέον να προωθήσει και τη συνεργασία με τα κράτη-μέλη στον τομέα αυτό. Υπάρχει κάποια κράτη-μέλη έχουν ορισμένε επιφυλάξεις, κάποιους φόβους για το κίνδυνο να χρειαστούν νέες επενδύσεις από αυτούς που έχουν ήδη προχωρήσει επενδύσεις ε, για νέα πρότυπα ή νέα, νέες εγκρίσεις τύπου. Είναι σημαντικό λοιπόν να υπάρξει μια νέα πλατφόρμα ενιαία ούτως ώστε τα κράτη-μέλη και όλοι οι ειδικοί να μπορούν να συναντηθούν για να συζητήσουν τα ζητήματα και ούτως ώστε ε, οι δράσεις και τα πρακτικά ε, έργα ε, να μπορέσουν να υλοποιηθούν σε ένα κοινό, ε, κοινώς αποδεκτό κλίμα. Δείξαμε στο ντοσί αυτό ότι είναι σημαντικό όχι μόνο να επιβάλλουμε εκ των άνωθεν λύσεις αλλά και έναν διάλογο εκ των κάτω. Θέλω να υπενθυμίσω επίσης ότι στο Κοινοβούλιο έγινε μια συζήτηση για τα ευφυΐ συστήματα μεταφορών καθιστούν για να δούμε αν μας κάνουν πιο έξυπνους ή πιο χαζούς. Αλλά και τα ευφυή συστήματα μεταφορών πρέπει να χρησιμοποιούνται με ευφυή τρόπο. Αυτό είναι η βάση της δικής μου παρέμβασης. Και το GPS από μόνο του δεν έχει νόημα αν δεν χρησιμοποιείται με ευφυή τρόπο. Όταν σου λέει πρέπει να πας αριστερά και εσύ πας δεξιά, τι ευφυές σύστημα να είναι αυτό. Ευχαριστώ. Κυρία Γένσεν, λέει ο ε, Uh, η συζήτηση ολοκληρώνεται και η ψηφοφορία θα λάβει χώρα, χώρα αύριο στις 12. Προχωρούμε τώρα στο επόμενο θέμα, η έκθεση Στέρξ για τις διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων πλοίων. Ο κύριος Στέρξ έχει το λόγο.